τι ομάδε ε, του ΕΛΚ, ε, των Σοσιαλιστών και Δημετρατών, ε, των Φιλελευθέρων και του EFTD κάποια αιτήματα για διορισμού σε επιτροπέ και σε μια αντιπροσωπεία. Αυτέ οι διορισμοί θα αναφέρονται στα πρακτικά αυτή τη συνεδρίαση και αν δεν υπάρξει παρατήρηση μέχρι την έγκριση των πρακτικών θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται και αυτοί οι διορισμοί. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, Γιούλια Πιτέρα, στη θέση του κυρίου Σάιρο Βόλσκι. Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, Μισάλ Μπόνι, στη θέση του Γιάρο Βόλσκι. Επιτροπή Αναφορών, Μάριος Βόλσκι στη θέση της Γιούλια Πιτέρα. Επιτροπή για την έρευνα για τις ε, παραβιάσεις σε θέματα εφαρμογής ε, του δικαίου της Ένωσης όσον αφορά την ομοιοποίηση παρανόμων εσόδων, φοροδιαφυγή και απορροφυγή. Βίρκο Νεγκρέστου στη θέση του Καταλίν Σόρινοβ Ήβαν αντιπροσωπεία για την Ελβετία και την Νορβηγία, η Μικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισλανδίας και τη ΕΟΧ Νίλ Στόρβα, αποσύρεται από τη θέση του. Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, ο κύριος Φίντς αντικαθιστά τον κύριο Έθεριτζ. Διάφορε αντιπροσωπείε αποφάσισαν να ξεκινήσουν διοργανικέ διαπραγματεύσει βάσει του άρθρου 69 Γ, παράγραφο 1 του